του πρώτου σημείου. Μάλλον πρώτα η έγκριση των χθεσινών πρακτικών. Λάβατε τα χθεσινά πρακτικά, ήθελα να ξέρω αν έχετε παρατηρήσεις. Δεν νομίζω ότι έχει